το εννοώ τέλος ε, βάσει του άρθρου 216 του εσωτερικού κανονισμού οι επιτροπές που είναι αρμόδιες για διάφορα διορθωτικά κείμενα ε, νομοθετικής φύσης που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο ε, πρώτον ε, συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών δείτε τα διορθωτικά σημειώματα υπάρχουν στους φακέλους σας κατόπιν κανονισμός του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ονοματολογία των ινών και επίσης τη θέση σε εμπορία, την παραγωγή και θέση σε εμπορία των κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων και εκεί υπάρχει ένα διορθωτικό σημείωμα, επίσης είναι στους φακέλους σας βάσει του άρθρου 216.4 τα διορθωτικά σημειώματα θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εκτός αν προβάλλεται ενστάσεις σε διάστημα 48 ώρων μετά τη δημοσίευσή τους και εκτός και αν ζητήσει μια πολιτική ομάδα, τουλάχιστον 40 μέλη, να γίνει ψηφοφορία. Επίση υπάρχουν επιγραμμικά στο, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου αυτά τα διορθωτικά σημειώματα. Φτάνουν στο τέλο των ανακοινώσεων και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη τη ε, Συνόδου. Έχετε την ε, τελική ημερήσια διάταξη που ενέκρινε η διάσκεψη των Προέδρων στι 7 ε, Σεπτεμβρίου και βάσει του άρθρου 137 του κανονισμού.